Περνάμε τώρα, μάλλον έχουμε έξι ψηφίσματα για την λήξη της συζήτησης. Τώρα θα λάβει χώρα αμέσως η ψηφοφορία των ψηφισμάτων. Ερχόμαστε πρώτα στην ψηφοφορία σε σχέση με την κατάσταση στην Καμπότζη και το Λάος. Έχουμε το κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων, τροπολογία 8, ε, 6, Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Γίνεται δεκτή. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Δεκτή. Τροπολογία 8 με ονομαστική παλικλήση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απολύπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απολύπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Καρμέ, έλεγχο για την τροπολογία υπαριθμών 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4 μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία, Δεκτή. Το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Έχει εγκριθεί εκπίπτουν όλα τα άλλα ψηφίσματα κατά συνέπεια. Ερχόμαστε στην, στα ψηφίσματα σε σχέση με τις εκλογές των Μπαγκλαντές. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο. Αρχίζεται η ψηφοφορία έλεγχο. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο επομένως δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Παράφος 9. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τέλος το ψήφισμα για τις νέες κινήσεις ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜΑ. Κύριε Σπότη, για διαδικαστικό θέμα. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε, και ο Σπόσελτ έχει παρουσιάσει ένα ψήφισμα η δική μου πολιτική ομάδα, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο κοινό ε, ψήφισμα αλλά δεν βρίσκεται στους φακέλους μας και δεν έχει μεταφραστεί. Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το συνηθισμένο. Όταν υπάρχουν κοινά ψηφίσματα τα αρχικά κείμενα δεν είναι πια διαθέσιμα. Μόνο όταν ένα τμήμα <clears throat> των κομμάτων έχει ένα κοινό ψήφισμα και τα άλλα δεν συμμετέχουν τότε θα πρέπει η Ολομέλεια αμφασίσει αν θα υποστηρίξει το κοινό ψήφισμα ή τα μεμονωμένα ψηφίσματα. Σας παρακαλώ στο μέλλον. Όταν δεν συμμετέχει μια πολιτική ομάδα στο κοινό ψήφισμα, το κείμενο αυτό να μεταφράζεται και να είναι διαθέσιμο και να είναι διαθέσιμο στους φακέλους των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ. Το λαμβάνουμε υπόψη. Εγώ πιστεύω ότι συμφωνώ, μαζί σας και θα πρέπει αυτό να γίνει δεκτό στην πρακτική μας όταν μια ομάδα δεν έχει υποστηρίξει ένα κοινό ψήφισμα ότι θα πρέπει το εναλλακτικό κείμενο να είναι στη διάθεση των βουλευτών στη μητρική τους γλώσσα. Αλλά, κύριε Πόσελτ, αυτός δεν είναι λόγος για να αναβληθεί η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν. σε ένα αρχικό κείμενο. Ψήφι ΠΕΡ. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω ότι εξεπλάγει και εγώ που ε, ε, δεν ε, βρήκα αυτό το ψήφισμα του ΕΛΚ παρότι δεν είχα καμία πρόθεση να το ψηφίσω. Εξεπλάγει. πραγματικά πρέπει να, έπρεπε να είναι παρόν στο φάκελό μας το κείμενο αυτό εφόσον ε, σα ενδιαφέρει αυτό, θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα σε το κείμενο αυτό να είναι στη διάθεση των βουλευτών. Παράγραφο ένα αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Δεκτή. Παράγραφος 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο για την παράγραφο 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την παράγραφο 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ. Άμα βγάλετε την κάρτα σας πριν από την, ε, το τέλος της ψηφοφορίας, τότε χάνετε η ψήφο σας. Παραφό 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος για τη 12 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 αρχικό κείμενο. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Κύριε Πρέντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Απλώς θέλουμε να προσθέσουμε στην παραγράφο 14 την Ρωσία όσον αφορά ε, τους, ε, δηλαδή να πούμε ε, τον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο της χώρας. Δεν είχαμε ξεχάσει, είχαμε ξεχάσει την Ρωσία στους αποδέκτες του ψηφίσματος. Έχετε αντιρρήσει την προφορική τροπολογία? Όχι. Λοιπόν, παράγραφος 15, το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ετιολογική σκέψη 7, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική σκέψη Β, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε τελειώσει κυρίες και κύριοι. Σας εύχομαι καλή επιστροφή στις αιστείες σας. και έχει τελειώσει η συνεδρίαση.